Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ladies and gentlemen, please be seated. Κυρίες και κύριοι, καθίστε σας παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ξεκινάμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της ε, υποεπιτροπής μας. Το μόνο ουσιαστικό σημείο που έχουμε στη Μέση Διάταξη είναι η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης με θέμα την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η SDP. Πρωτού προχωρήσουμε όμως στην ε, συζήτηση, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όπως πάντοτε η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και όσον αφορά τη διερμηνία, προτεραιότητα δίνεται στις γλώσσες των τακτικών μελών της υποεπιτροπής μας. Λόγω της ειδική διαδικασία που θα ακολουθηθεί σήμερα στη συνεδρίαση όμως, δυστυχώς πρέπει να σας ανακοινώσω ότι δεν υπάρχει διερμηνία στα τσεχικά και στα κροατικά. Α, έχουμε. Α, με συγχωρείτε, τότε άλλαξε. I long trip, uh, just... Συγγνώμη, ε, μόλις ήρθα από το αεροπλάνο Είχα μεγάλο ταξάδιο, ταξίδι, δεν είχα δει αυτή την αλλαγή. Σας ευχαριστώ παρόλα, αυτό, ε, παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς και την γραμματεία που εξασφάλισε τη διερμηνία και σε αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι τη Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, στην ε, Ολομέλεια στο Στρασβούργο, στις 7 το βράδυ, θα γίνει διευρυμένο προεδρείο όπου θα ε, εξεταστεί το ζήτημα των υπολοιπόμενων ακροάσεων, άλλων δραστηριοτήτων που έχουμε προγραμματίσει, κάποια άλλα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν ως υποεπιτροπή μέχρι το τέλος της θητείας και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συντονιστές να παρευρεθούν σε αυτήν τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο επίγον ζήτημα που χρειάζεται να σας ε, ανακοινώσω και γι' αυτό χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας τον κύριο Μιτσέα Πάσκου και θα ανακοινώσω, θα τα πω όλα και μετά την ε, τοποθέτησή του Απλά να σας πω από τώρα ότι έχει πάρει παράταση η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Είναι πλέον στις 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι η προθεσμία αυτή. Έως εκείνη την ημερομηνία και ώρα μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Κύριε Πάσκου, έχετε το λόγο. sorry. I would like to... Συγγνώμη. Θα ήθελα επίσης θερμότατα να καλωσορίσω τα μέλη του Σεμιναρίου Υψηλού Επιπέδου για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας που συμμετέχουν σήμερα εδώ στη συνεδρίασή μας και να ανακοινώσω ότι μετά την έκτακτη συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ θα γίνει συνάντηση με τα μέλη αυτού του Σεμιναρίου Υψηλού Επιπέδου. Ε, Van Orden, would you like... Κύριε Βανόρντεν, θέλετε να πείτε κάτι?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 right, I will speak uh, Εντάξει, θα μιλήσω αγγλικά αφού δεν υπάρχει διερμηνία. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν μια σειρά από κεφάλαια, τίτλους. Το πρώτο αφορά το ε, στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης, το οποίο επιδεινώνεται και γνωρίζουμε όλοι την σειρά απειλών, κινδύνων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Κατά τη γνώμη μου όμως, αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική πρόσκληση, πρόκληση. Το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες για τη διεθνή τάξη βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Το ελεύθερο εμπόριο αμφισβητείται και γι' αυτό το λόγο Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί συστατικό στοιχείο του γενετικού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελεύθερο εμπόριο, οι ελεύθερες συναλλαγές αποτελούν τον εγκέφαλο, τον βασικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, ε, αντιμετωπίζει συστημική πρόκληση. Πέρα από τις ε, ε, φυσικές καταστροφές, την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις μεταξύ κροτών, τις ε, υβριδικές απειλές κτλ. κτλ. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή είναι η, βασική ε, προσθήκη όσον αφορά την αξιολόγηση. Μετά υπάρχει ένας τίτλος σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα στην κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας. Πρέπει να γίνουν ε, οι κατάλληλες και ε, ενδεικνυόμενες ε, επενδύσεις υπό τις περιστάσεις που βρισκόμαστε και αυτό συνάδει και με την, την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και η παράγραφος 8 που είναι πολύ σημαντική διότι υπάρχουν, έχουν ήδη ληφθεί μια σειρά από διαχειριστικά μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα υπάρχει πλέον ε, αντίστοιχο κεφάλαιο και στην πρόταση της ε, Κομισιόν για, την, για το ΠΔΠ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια γραμμή ε, από την, του προπολογισμού από την οποία θα χρηματοδοτούνται έργα που θα αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα. Μέχρι σήμερα ε, ο κλάδος αυτός, ο τομέας αυτός βρισκόταν διασπαρμένος σε διάφορες γενικές διευθύνσεις. Πλέον έχουμε μία γραμμή, έναν τίτλο και το λογικό συμπέρασμα, η λογική συνέπεια θα ήταν να προσαρμοστούμε και να, ε, να ζητήσουμε και μια κεντρική διαχείριση σε επίπεδο Επιτροπής των ζητημάτων που σχετίζονται με την άμυνα. Επίσης, Υπάρχουν μια σειρά από έργα. Το, στο, στο EDF, το Ταμείο για την Άμυνα, υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες αναφορές και την ιεράρχηση των έργων αυτών. Όταν κανείς ζητά χρήματα για συγκεκριμένα έργα ή και, συνδέει τα έργα αυτά με την αξιολόγηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την, την, την τήρηση αυτών σε, κάποιο, σε κάποια χώρα, αυτό είναι πράγματι ένα θέμα. Δεύτερον όμως, η ασφάλεια έχει έναν, ε, ε, έχει έναν χαρακτήρα αδιέρετο. Δεν σχετίζεται με το, με το ποια είναι η, εκτίμησή μας για το αν και κατά πόσο εφαρμόζεται η... ο νόμος και η τάξη σε μια χώρα. Ξέρετε όμως πώς ε, συζητιούνται αυτά τα θέματα. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα έχουμε μια καλή ευκαιρία να δούμε αυτή... αυτή την αυτών των, των, τη συνεκτίμηση όλων αυτών των διαστάσεων. Πρέπει λοιπόν να ε, αποφύγουμε πάση θυσία την πολιτικοποίηση αυτής της συζήτησης. Επίσης, επαναφέρω την ιδέα της Λευκής Βίβλου. Ξέρετε ότι αποτελεί πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου η σύνταξη μιας τέτοιας Λευκής Βίβλου προς εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ε, λήψη της σχετικής απόφασης. Επίσης, ικανότητες για την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης. Είναι και αυτό ένα θέμα της ετήσιας έκθεσης. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλα όσα κάνει ένα κράτος μέλος όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα ε, ενισχύει και το ΝΑΤΟ. Ενισχύουν και το ΝΑΤΟ. Ακόμη και αν δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ενισχύεται η κοινή ασφάλεια και άμυνα στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε αυτό τον τομέα και υπάρχει και μια παράγραφος, η παριθμόν 15, που είναι τροφή για σκέψη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όλα όσα έχουμε, να τα κεφαλαιοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα και να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα για να μπορέσουμε να συνενώσουμε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία που έχουμε για να ε, ε, καθορίσουμε και να καταρτήσουμε, να χαράξουμε μια μελλοντική πολιτική. Μετά υπάρχει το EDIDP, ε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αμυντική Βιομηχανία, υπάρχει η παράγραφος 20 που αφορά το EDA, που είναι μια πρωτοβουλία διακρατική να μην ξεχνούμε όμως ότι υπάρχει μια συσσόρευση εμπειρίας, τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης ε, στο EDA που δίνει τη δυνατότητα στο φορέα αυτό να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας, των συμπράξεων μεταξύ των κρατών. Επίσης, Υπάρχουν οι αποστολέ τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, οι αντίστοιχε επιχειρήσει. Αναφέρονται όλα αυτά ε, μέσα στην έκθεση προσπαθούμε να καταγράψουμε το πού βρισκόμαστε και υπάρχει και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι συμπληρωματική η συνεργασία, να λαμβάνει υπόψη τις, ε, τους, ε, τις ιδιαιτερότητες ε, και τους ρόλους του καθενός, κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επί μακρόν και με άλλες ευκαιρίες. Επίσης, ε, εκφράζεται υποστήριξη στη διακήρυξη των Βρυξελών, για την υποστήριξη των προσπαθειών για την στρατιωτική κινητικότητα και ε, αναφορά στο ότι η ΠΕΣΚΟ είναι συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ. Νέο, νέο κεφάλαιο είναι οι εταιρικέ σχέσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε πάντοτε να κάνουμε με τα ίδια ακριβώ μέλη των, των, των οργανώσεων, αλλά και με χώρες που συμμερίζονται τις αξίες μας και τις αρχές μας, αλλά όχι μόνο χώρες και φορείς. Υπάρχουν λοιπόν δύο ε, παράγραφοι οι οποίες είναι αφιερωμένες σε αυτό ακριβώς το θέμα, την ε, συμμετοχή, την ε, συνεργασία με τους εταίρους μας. Και υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αφορά την κοινοβουλευτική διάσταση. Ξέρετε ότι όσο περισσότερα χρήματα κατευθύνονται στην ασφάλεια και την άμυνα, τόσο μεγαλύτερο έλεγχο θα πρέπει να ασκεί το κοινοβούλιο σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι αναπόφευκτο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η λογική συνέπεια όλων αυτών είναι να εξετάσουμε για άλλη μια φορά σοβαρά ε, να ε, προάγουμε την υποεπιτροπή μας στο καθεστώς μιας πλήρους επιτροπής. Με αυτά ολοκληρώνω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πάσκου. Uh, Ο κύριος Στανσόν είναι σκιώδης για το ΕΛΚ. Ε, Αποουσιάζει όμως. Δεν μπόρεσε να έρθει στις Βρυξέλλες για αυτή τη συνάντησή μας. Ο κύριος Μιχαλ Κάλερ θα μιλήσει εκ μέρους του ναι, όντως πρώτα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ο κύριος Στανίσα στα συγγνώμη για την απουσία του. Ευχαριστεί τον εισηγητή για τη θαυμάσια εργασία. Η έκθεση αυτή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση και καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της άμενας της Ένωσης καθώς και της ανάπτυξης της στρατιωτικής δυνατότητας της Ένωσης. Έχουμε και κάποιες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την ενίσχυση της έκθεσης. Και ήδη αναφερθήκατε στην αναβάθμιση της Επιτροπής, κάτι το οποίο συμμερίζομαι και εγώ. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιμένουμε ώστε και η Κομισιό να δημιουργήσει αντίστοιχα μια γενική διευθυνσία άμυνας, DG Defense ή κάτι αντίστοιχο Τώρα υπάρχουν αρκετά κονδύλια και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και σε επίπεδο διοικητικό στην Κομισιόν αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε λοιπόν και στηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ECR. Ο κύριο Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή του έκθεση, η οποία επί το πλήστο όμως με βρίσκει αντίθετο. Αυτό που εξέφρασε στην αρχή της ομιλίας σου, κλάτε και στο προήμιο της έκθεσης με τα νέα αυτά στοιχεία και βεβαίως αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για μας ως βουλευτές ε, να πούμε τα πράγματα ως έχουν, όχι ζώντας ένα φανταστικό κόσμο. Δεν είμαι βέβαιος λοιπόν ότι το στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης είναι διαφορετικό από το στρατηγικό περιβάλλον του ΝΑΤΟ ας πούμε. Ακούμε πολλά και για την Αφρική. Ξέρω ότι υπάρχει μια ειδική σχέση των Γάλλων με την Αφρική και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται από αυτό. Παρ' όλα αυτά, Έχουμε και την κλίμακα της ανάμεξης άλλων χωρών στην Αφρική, η οποία είναι πολύ ψηλότερη από αυτή των χωρών της Ένωσης, όπως ας πούμε η ΕΠΑ. Έχουν 68 επιχειρήσεις, τουλάχιστον κοινέ επιχειρήσεις επίσης, μορφές συνεργασίας, εκατοντάδες, έχουν επενδύσεις, και πολλές άλλες δραστηριότητες στην Αφρική οι Αμερικανοί. Υπάρχει λοιπόν τεράστια συμμετοχή, η παρουσία των ΗΠΑ στην Αφρική. Δεν είναι μόνο αρμοδιότητα η ευθύνη της Ένωσης αυτό, όπως θεωρούν κάποιοι. Και άλλες χώρες, όπως και η Κίνα είναι παρουσίες, όπως η Ινδία και αυτές στην Αφρική. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα σχέση με το στρατηγικό περιβάλλον. Εσείς Αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όχι με τη σωστή προσέγγιση. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί λογικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υπερασπιστεί την Ένωση είτε τώρα είτε στο μέλλον. Βασιζόμαστε στις ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ και στις, εξυγχρονι... στις σύγχρονες δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις των χωρών μας. Αυτό κάνουμε στην Ευρώπη και αυτό θα αποτελέσει μια αξιόπιστη αποτροπή προς τον Πούτιν και άλλους επίδοξους. Δεν αναφέρεστε καθόλου στο Brexit μάλιστα. Ξέρω ότι κάποιοι μάλιστα δίνουν ιδιαίτερη σημασία όπως εμείς οι Βρετανοί. Βεβαίως θα θέλαμε να έχουμε μια ισχυρή σχέση με την Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Αφού το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το μεγαλύτερο συμβάλλοντα στην Ένωση όσον αφορά το στρατιωτικό δυναμικό και την εμβέλειά του και μιας και θα χαθεί πέρα από το προπολισμό θα χαθεί και αυτό το στρατιωτικό στοιχείο. Ακούσαμε αυτέ τι ωραίε ιδέε για τα νέα χρήματα και νέα κονδύλια που θα δαπανηθούν. Να θυμάστε όμω ότι το Ηνωμένο Βασιλείο είναι ο δεύτερο ε, συνεισφέροντα στον προπολογισμό τη Ένωση. Δηλαδή δεν γίνεται οι Γερμανοί μέσω των φορολογουμένων τους να συνεχίσουν να διασώζουν τους υπόλοιπου. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιον ρεαλισμό εδώ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή την ενωσιακή στρατηγική αυτονομία. Άλλη μια γαλλική ιδέα αυτή. Τι σημαίνει αυτό. Στρατηγική αυτονομία σημαίνει απουσία τον ΗΠΑ, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Ναι, ναι, αλλά δεν το προσδιορίζεται. Το αναφέρετε, το αναφέρετε, εντάξει, το αναφέρετε. Αλλά δεν το προσδιορίζετε και δεν ξέρει κανείς τι εννοούμε εδώ και αυτό είναι επικίνδυνο έννοια. Πάντως ανησυχώ σε σχέση με αυτή την επικάλυψη δομών και την ε, παρέκκληση πνευματικής προσπάθειας που θα πάει σε αυτό το εγχείρημα τη στιγμή που χρειαζόμαστε μία αναθέρμανση της σχέσης μας με το ΝΑΤΟ ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και καμιά από τις αποστολές της Ένωσης δεν αντέχουν σύγκρισης. Αν δείτε και την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου λένε ότι αυτές οι αποστολές της Ένωσης εμφανισιακά είναι πολύ ωραίες, αλλά η πραγματικότητα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι τελείως διαφορετική. Οπότε νομίζω ότι εδώ πραγματικά χάσατε την ευκαιρία στην έκθεση να δείξετε περισσότερο ρεαλισμό για το πού ακριβώ βρισκόμαστε. Αυτά που ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ζωράντος είναι εκείνος που θα εκπροσωπούσε τους φιλελεύθερους, αλλά δεν είναι εδώ ούτε εκείνος. Λόιζινγκ απουσιάζει επίσης. Η κυρία την Βαλέρο, λοιπόν, σκιώδης συγκήτρια για τους πράσινους. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ειδικά, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Πάσκου για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν συμφωνούμε πάντοτε μεταξύ μας. Όμως μετά από διάφορες συζητήσεις με τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις καταφέραμε να πετύχουμε κάποιες συγκλήσεις. Να ξεκινήσω με τα θετικά στοιχεία της έκθεσης. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια εναλλακτική. Η μόνη δυνατότητα, η μόνη επιλογή είναι η συνεργασία, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά ασφάλεια. Και μετά συμφωνώ για τι αλλαγέ τη δομική που πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μ' αρέσει επίση το τμήμα τη έκθεση όπου γίνεται λόγο για αυτό το peace facility στην παράγραφο 12. σω όμω να πρέπει να αλλάξουμε την ορολογία, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την ειρήνη, την οικοδόμηση ειρήνη, αλλά την διατήρηση της ειρήνης με κάποιες επιχειρήσεις. Οπότε αυτό το facility, αυτή η δομή θα πρέπει να έχει διαφορετικό όνομα. Παράγραφος 15. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, γιατί θα ήταν απαραίτητο κατά την άποψή μου να έχουμε μία πολυεθνική δομή σε μόνιμη βάση. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα θα αναφερθώ στα αρνητικά, στα σημεία που με βρίσκουν αντίθετη. Ένα από τα κυριότερα είναι οι προτάσεις για τα κονδύλια της Ένωσης που αποσκοπούν στη χρήση για τις στρατιωτικές δομές και τις επιχειρήσεις ασφάλειας. Όμως με τις προτάσεις αυτές παραβιάζουμε νομίζω τη συνθήκη. Εμείς πρέπει να τηρούμε τους δικούς μας κανόνες. Γιατί θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτές οι δαπάνες να βαραίνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Τώρα για τις στρατιωτικές δομές και υποδομές. Μιλάμε κυρίως για το ΝΑΤΟ. Αλλά αυτή η μορφή άμυνας νομίζω ότι δεν αφορά ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και τον εξάρτητο ΝΑΤΟ. Μετά παράγραφος 18, το Ταμείο για την Άμυνα. Να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπα προηγουμένως, ως σημείο κίνησης, δηλαδή ότι τα όπλα δεν θα πρέπει να αγοράζονται οι εξοπλισμοί, δηλαδή θα πρέπει να γίνονται μέσω αυτού του ταμείου. Γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνά είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορεί όμω να αποτελέσει μια λευκή επιταγή για να, κάνει, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μετά, όταν μιλάμε για αυτή την υπηρεσία άμυνα, έχουν περάσει 15 χρόνια με προσπάθειες που έγιναν για βελτιώσεις, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Οπότε η Κομισιόν τώρα θα πρέπει να προσπαθήσει να συνεργαστούν με τρόπο αποτελεσματικό οι χώρες μέλη, ώστε ακριβώς να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, να αποφύγουμε τους κατακαιρματισμούς, να αποφύγουμε αυτή την ε, βιομηχανική υπερεκμετάλλευση. Τώρα, κάποια άλλα σχόλια. Γενικότερα ίσως. Εδώ στην έκθεση μιλάμε κυρίω για στρατιωτικές παρεμβάσεις. Όμως, αν κοιτάξουμε τις δικέ μας ε, παρεμβάσεις, αυτές οι παρεμβάσεις έχουν κυρίω πολιτικό χαρακτήρα και όχι κυρίω στρατιωτικό. Οπότε θα έπρεπε στην έκθεση να επικεντρωθούμε και σε αυτές τις πολιτικές μας παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ανέλη. ευχαριστώ πολύ Γεια σας. Ε, θα ήθελα ε, να αναφερθώ κι εγώ ε, στην πρώτη αυτή παρουσίαση. Σε σχέση με αυτό που υπόθηκε προηγουμένω από τον κύριο Φανόρδο, ναι, η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορώ να σα δώσω πολλά παραδείγματα ε, προ ε, την κατεύθυνση αυτή. Ε, Καταρχά, πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει μια συγκέντρωση πόρων από του οποίου μετά θα αντλούμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που μπορούμε να συγκεντρώσουμε ω πόρου. Η αυτονομία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι μια διπλή δομή ή είναι ε, επίσης το κομμάτι που αφορά καθαρά ε, και τον κυβερνοχώρο και τη σχέση με το στρατιωτικό τομέα, πώς είναι δυνατόν να ορίσουμε αυτήν την ε, ικανότητα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της αυτονομίας. Θα μπορούσαμε ίσως αυτό το κομμάτι του κυβερνοχώρου να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση, ότι έχει ενισχυθεί δηλαδή ε, υπήρξαν ήδη κάποιες νήξεις ε, προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάει αυτό το ζήτημα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι η ραχοκοκαλιά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ε, η συγκέντρωση πόρων αλλά και η άντληση στη συνέχεια από αυτούς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να την χάνει κοινοβουλευτικής εξέτασης και ακριβώς αυτό ήθελε να πει και η κυρία Βαλέρο όταν έλεγε ότι πρέπει να ξέρουμε σε τι ξοδεύουμε τα χρήματα. Υπήρξε μάλιστα και μία ερώτηση προς τη γερμανική κυβέρνηση όταν ε, ακούστηκε ότι δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ ε, όταν δεν υπάρχουν ε, προγράμματα γερμανικής προέλευσης, όμως δεν ισχύει πάντοτε αυτό. Η ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα. Ε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω να το ε, ξανασκεφτούμε, να σκεφτούμε η δική μας επιτροπή να γίνει πλήρης επιτροπή και όχι να παραμείνει υποεπιτροπή, γιατί έτσι θα είμαστε και πιο ορατοί νομίζω ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, θα μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε και σε επίπεδο κρατών μελών ε, για να μπορούμε να έχουμε και την ευκαιρία να αποφασίζουμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Κατά γνώμη μου έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεση. Ε, και ένα τελευταίο Αναφέρατε το Brexit. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναφέρεται. Βέβαια δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Είδαμε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά νομίζω ότι κάπου θα έπρεπε να το αναφέρουμε. Ίσως όχι λεπτομερός. Να... Είναι μια κατάσταση την οποία την προβλέπουμε εν πάση περιπτώσει και τη λαμβάνουμε υπόψη ε, χωρίς να μπούμε σε πάρα πολύ λεπτομέρεια. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί ε, ίσως μέσα μέσω του Brexit καταφέραμε να μιλήσουμε επιτέλους για αυτήν την ευρωπαϊκή αυτονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία που είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση και είναι και πολύ σημαντική. και δείχνει ότι υπάρχει μια αλλαγή πολιτική ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Τονίζεται μία ακόμη φορά στο έγγραφο αυτό ότι τα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας ε, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, έχουν, αποτελούν πλέον το επίκεντρο της προσοχής εγώ δεν είμαι πάρα πολύ πεπισμένος από όλες αυτές ε, τις ε, επιφυλακτικές και σκεπτικιστικές φωνές που ακούγονται. Κατά τη γνώμη μου αποδυναμώνουν ε, τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι στο έγγραφο αυτό τονίζεται πολλές φορές ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ θα παραμείνει μεγάλη σημασία, ζωτική σημασία, επειδή υπάρχουν και προσδοκίε ε, και από πλευρά ε, Ηνωμένων Πολιτειών προ τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε όλα αυτά τα ε, στοιχεία που οδηγούν σε μια κάποια αυτονομία. Θα ήθελα να τονίσω τα εξή σημεία τα οποία ε, τόνισε και ο εισηγητής στην έκθεσή του. Καταρχάς, ε, την, ε, τη στρατιωτική ικανότητα. Δεύτερον, την ε, λευκή βίβλο στην οποία αναφερθήκατε και την παρακολούθηση, δηλαδή μέσω της παρακολούθησης θα μπορούσαμε να, ξέραμε καλύτερα, να ξέρουμε καλύτερα ποια είναι η κατάσταση των ρυθμικών μας δυνάμεων, της επιμελητίας μας και θα μπορούσαμε ε, ταχύτερα να ανταποκρινόμαστε ε, σε διάφορα προβλήματα που ενδεχομένως να έχουμε και να αντιμετωπίσουμε κάποιες αδυναμίες μας. Επίσης πρέπει να αναβαθμίσουμε την υποεπιτροπή μας, να αποτελεί πλέον μία πλήρη επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών μας. Ε, η Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας ε, να αναβαθμιστεί σε πλήρη επιτροπή. Τώρα, το τρίτο σημείο, το Brexit ε, υπάρχει μια αλλαγή της κοινή γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αν τη λάβουμε αυτήν υπόψη πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή αναστάτωση και διακοπή ε, σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, η ασφάλεια και η άμυνα σημαίνουν ε, ε, ασφάλεια και του στρατιωτικού τομέα αλλά και των πολιτών. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή αναστάτωση μεταξύ των, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στετίνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τσέχικα. Καλησπέρα. Κύριε Πάσκο, σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Κατανοώ όλα αυτά που είπατε. Όμως υπάρχει ε, κάτι που λείπει. Ένα κεφάλαιο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που λείπει. Στην υποεπιτροπή μας την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνα, έχουμε πολύ συχνά προσκεκλημένου εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και σε μια σειρά από περιπτώσει έχουμε συζητήσει ε, ζητήματα που σχετίζονται με απειλές και κινδύνους στην ασφάλεια. Απειλές ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα κράτη-μέλη. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι μήπως θα πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτές τις απειλές εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο. Μήπως θα έπρεπε να γίνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένε απειλές και κινδύνους που πηγάζουν από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα ήθελα επίσης να γίνει μεγαλύτερος λόγος ε, σχετικά με το άρθρο 5 και την εφαρμογή του, του χάρτη του ΝΑΤΟ για την αλληλοβοήθεια που προσφέρουν τα μέλη του ΝΑΤΟ το ένα στο άλλο σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεχτεί επίθεση. Ποτέ όμως δεν έχει αναφερθεί ρητός τι θα συμβεί σε περίπτωση που μία από τις βαλτικές χώρες δεχτεί επίθεση όπως η επίθεση που έγινε από τους πράσινους στρατιώτες. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία, συγκεκριμένη κατεύθυνση και απόφαση για το τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που επέλθει μια τέτοια κατάσταση και δεχτεί κάποιος επίθεση πραγματική. σε ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να παρέμβω ως μέλος της Επιτροπής μας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκο για την έκθεσή του Νομίζω ότι αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τη συζήτηση που θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία μέσω των συντονιστών για την τελική μορφή της έκθεσης για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, στρατηγική αυτονομία. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε σχέση με αυτήν την έννοια. Ε, στην πραγματικότητα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει σαφής ορισμός των τομέων στους οποίους είναι εφικτή μια στρατηγική αυτονομία και δυνητικά ωφέλιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιους τομείς ενδέχεται να ενέχονται κίνδυνοι από τη στρατηγική αυτονομία. Συμφωνώ με τον κύριο Βαν ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα των Αμερικανών είναι ύψιστη σημασία για την ασφάλεια της Επίρου μας και αύριο μεθαύριο όταν θα αυξηθούν και οι δαπάνες στην κατεύθυνση της κοινή άμυνας τότε μπορεί και να εξετάσουμε ε, σοβαρότερα το θέμα της κοινή μας άμυνας και της αυτονομία μας. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ επιφυλακτική υπό τις παρούσες, ε, υπό τις παρούσες περιστάσεις και συνθήκες. Τώρα, όσον αφορά την αναβάθμιση ε, και συγγνώμη που ξεκινώ έτσι άμεσα και, και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Έχω, είμαι, ε, είμαι άγρυπνη από τις 3 το, το, το, το πρωί. Τα ξημερώματα ξεκίνησα το, το ταξίδι μου. Ελπίζω να τα καταφέρω να το βγάλω το απόγευμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια, σε σχέση με την αναβάθμιση τη Επιτροπή μα, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Θεωρώ ότι τα ζητήματα ασφάλειας σχετίζονται στενά και αλληλοσυνδέονται με, με τις εξωτερικές υποθέσεις. δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει ολοκληρωμένα ε, την άμυνα, την ασφάλεια ενό ενός παγκόσμιου παίκτη όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν συνεκτιμήσει και δεν λάβει υπόψη, του, υπόψη και εξωτερικούς παράγοντες τις συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη γειτονία μας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα από μια τέτοια αναβάθμιση γιατί αυτή τη στιγμή η σύνδεσή μας με την ΑΦΕΤ, με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφτούμε για παράδειγμα την Ανατολική Ουκρανία Πήγαμε για παράδειγμα πρόσφατα στη Μαριούπολη, στην, ε, στις ακτές της Ουκρανίας και είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε επιτόπου την κατάσταση της ασφάλειας εκεί. Άρα θέλω να πω ότι οι δραστηριότητες μας αυτή τη στιγμή δεν αφορούν μόνο την παρακολούθηση των ε, μέτρων εφαρμογής της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αλλά προσπαθούμε να επικεντρωνόμαστε σε όλες τις παγκόσμιες απειλές και τους κινδύνους όπου και αν αυτοί εμφανίζονται. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει και μια πολύ θετική διάσταση ε, Αυτή τη σχέση μας με την ΑΦΕΤ. Αν από την άλλη μεριά η ΣΕΝΤΕ γίνει πλήρης επιτροπή, προφανώς ε, θα, θα τονιστεί βεβαίω η κοινοτική διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Αυτό είναι αλήθεια. Και για κάτι τέτοιο βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση και σύμφωνη γνώμη και των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν έχουν να παίξουν ρόλο και τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Και όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς λοιπόν θα ενισχυθεί η κοινωτική διάσταση από μια τέτοια αναβάθμιση ε, και εδώ πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Θέλουμε πράγματι κάτι τέτοιο ή όχι. Λοιπόν, δυστυχώς εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν έχουμε για να του δώσουμε το λόγο. Οπότε θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πάσκο για άλλη μια φορά για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις προτάσεις. Ξέρετε ότι ήταν αναπόφευκτο να απαντήσουμε στα πάντα από αυτή την πρώτη εκδοχή του κειμένου. Και άλλωστε σκοπός της σημερινής μας συζήτησης ήταν ακριβώς να ανοιχνεύσουμε τομείς που, να, που μπορούμε να ενισχύσουμε, να τους βελτιώσουμε, να μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αν θέλετε, να τους εξειδικεύσουμε περισσότερο. Από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρώ Τζόφρι Βαν Όρντεν ότι έχετε δίκιο. Ξέρετε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα συνεχιστούν οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανία στον τομέα τη άμυνα και τη ασφάλεια. Ενώ, όχι, εννοώ ότι δεν έχουμε ακόμα την τελική συμφωνία, δεν ξέρουμε πώ ακριβώ θα εφαρμοστεί, πώ θα υλοποιηθεί αυτά. Νομίζω παρόλα αυτά όμω ότι μπορούμε να καθορίσουμε κάποιε πολύ συγκεκριμένε αρχέ. Και να πούμε ότι επί της αρχής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί επί τόπου, να βασιστούμε σε αυτήν τη γνώση, σε αυτή τη χαρτογράφηση και την καταγραφή, αν θέλετε, της ίδιας της κατάστασης που επικρατεί και να βελτιώσουμε και να οικοδομήσουμε την περαιτέρω σχέση μας. Όσον αφορά τις ειδικέ επιχειρήσεις στην Αφρική, Πράγματι, ε, ενδεχομένως χρειάζεται μια αναφορά. Βλέπετε όμως ότι ακόμη και η Γερμανίδα Καγκελάριος ε, επισκέπτεται, επισκέφτηκε πρόσφατα την Αφρική. Όλοι αναφέρονται στην Αφρική, γιατί η Αφρική τα επόμενα χρόνια θα είναι μεγάλη πηγή προβλημάτων. Όπως και να έχει, η Αφρική ε, έχει ειδική θέση, έχει ειδικό ρόλο και συμφωνώ ότι Πρέπει να τονιστεί αυτό και στην έκθεση, να δοθεί δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στην Αφρική. Είπατε επίση ότι οι ΙΠΑ κάνουν περισσότερα από εμά. Ε, μα οι ΙΠΑ κάνουν παντού περισσότερα από εμά. Αν, αν, αν, είναι, ε, αν είναι να το πούμε αυτό, δεν, νομίζω ότι, ότι λέμε κάτι ιδιαίτερα ουσιώδες. Ξέρω ότι δεν, δεν εννοούσατε αυτό, απλά το, το τράβηξα λίγο στα άκρα για να, δω, για να σας δείξω τι, ποια είναι η δική μου στάση. Όπω και να έχει, όσα και να κάνει, περιθώρια βελτίωση και ενίσχυση των προσπαθειών υπάρχουν πάντοτε. Και με αυτό θέλω να έρθω στο θέμα τη ε, στρατηγική αυτονομία, την οποία απέφυγα σκοπίμω, γιατί ε, Αλλιώ ξεκινάμε, μια συζήτηση που δεν ξέρω αν θέλουμε να την κάνουμε. Τι είναι η στρατηγική ε, ε, αυτονομία, για παράδειγμα. Ο καθένα μπορεί να την ερμηνεύει διαφορετικά. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να μείνουμε εκτό αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια. Έχει κάνει πάρα πολλά σε σχέση με αυτό το θέμα. Σύνορα, ξέρετε τώρα. Ξέρετε, ξέρω ότι εσεί είστε απεσιόδοξο σε αυτά τα θέματα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Από μία άποψη λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια είναι ενισχυμένες και τείνουν να συγχωνευτούν και με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την εξωτερική ασφάλεια, ναι, πράγματι θα μπορούσε κανείς να εμπαράνει ότι αυτό είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αν θέλετε, αυτή τη έννοια στρατηγικής αυτονομίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα κίνδυνο. Ο κύριος Στέτινα αναφέρθηκε στο άρθρο 5. Νομίζω ότι ε, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος μιας έκθεσης για να θέσουμε ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 5. Αν ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε ε, σε έναν τομέα αρμοδιότητας που δεν είναι δικός μας, δηλαδή το άρθρο 5 δεν αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας με άμεσο τρόπο. Πάντως, δεν είναι καθόλου απίθανο να, ε, στο, στο, επόμενο διάστημα, στο μέλλον, να ενεργοποιηθεί ε, το, το άρθρο 5. Επίσης, ε, γίνεται μια δημόσια συζήτηση, εκτενής μάλιστα, για το Ποιο έχει δικαίωμα να το ενεργοποιήσει. Πόσο συμβάλλει κανεί στον προπολογισμό ε, του ΝΑΤΟ. Πόσο όχι. Πόσο συνδέεται αυτό με το δικαίωμα μια χώρα να ενεργοποιήσει το, το, ή να το επικαλεστεί το άρθρο 5. Υπάρχει επίση και το άρθρο 42 παράγραφο 7, το οποίο είναι ε, τελείω διαφορετικό θέμα πάλι και αποκαλύπτεται από άλλε εκθέσει. Λοιπόν, Αφρική, Brexit, σχέση με τη Βρετανία εν γέννη. Όλα αυτά πράγματι πρέπει να τα εξειδικεύσουμε περισσότερο, να τα ενισχύσουμε στην έκθεση. Περιμένω και τις τροπολογίες σας, αλήθεια, γιατί μέσα από αυτές τις τροπολογίες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε και σε συμβαστικές, αν θέλετε, λύσεις. Μη στρατιωτικό σκέλος των θεμάτων δεν έχει τονιστεί αρκετά. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση και προσοχή στα μη στρατιωτικά θέματα. Κυβερνοασφάλεια. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν, δεν, δεν εξειδίκευσα πολύ την κυβερνοασφάλεια γιατί δεν ήθελα να δώσω την, την εικόνα ή την εντύπωση ότι είναι σημαντικότερη από την κατεξοχήν ασφάλεια. Αλλά παρόλα αυτά, συμφωνώ μαζί σα ότι είναι σημαντικό να τονιστεί το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας ακριβώς γιατί διασυνδέεται με όλες τις διαστάσεις και τους τομείς της κατεξοχήν ασφάλειας. Υπάρχει μία απόκληση επίσης και μία αναντιστοιχία αν θέλετε μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Εμείς όμως είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και γι' αυτό είπα ότι όσο περισσότερη έμφαση δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ασφάλεια και στην άμυνα, τόσο περισσότερα χρήματα θα κατευθύνονται και τόσο, είναι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάγκη για, για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς αυτό κάνει άλλωστε. Ήδη στο επόμενο την δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνεται να κατευθυνθούν δισεκατομμύρια στον, ε, στον ενωσιακό προπολογισμό για την άμυνα. Δεν ήταν δική μου ιδέα όλα αυτά. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, τα προγράμματα για τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας κτλ. Κυρία Φωτίγκα. Γνωρίζετε ότι τα χρήματα για την παρότρινση και την ενίσχυση της ε, συνεργασίας στο ΜΕΤΣ Άμυνας ε, ε, είναι κάπως διάσπαρτα. Υπάρχουν διάφορε γενικέ διευθύνσει, διάφορα τμήματα, μονάδε κτλ, κτλ. που όλοι λίγο πολύ ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα της άμυνα και της ασφάλειας. Αν όμως συγχωνεύσουμε και εξορθολογήσουμε την χρήση όλων αυτών των κονδυλίων νομίζω ότι η λογική συνέπεια είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κέντρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κομισιόν. Εγώ δεν θέλω να, να το τραβήξω στα άκρα και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτό. Τα κράτη-μέλη στο κάτω-κάτω θα τα, θα τα αποφασίσουν όλα αυτά. Αλλά λέω ότι είναι η λογική συνέπεια του αιτήματο και των ετοιμάτων εν γέννη της δικής μας υποεπιτροπής. Αν γίνουν δεκτά αυτά που ζητάμε, είναι προφανές ότι θα, επιταχυνθούν, θα επιταχυνθεί μια τέτοια διαδικασία σε επίπεδο κομισιών. Εγώ δεν, δεν θα μπω στην ε, διαδικασία να υποβάλω συγκεκριμένες ε, προτάσεις, γι' αυτό και δεν έχω εντάξει κάτι τέτοιο στην έκθεσή μου. Εν περιπτώσει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε την προθεσμία στι 15 Οκτωβρίου για τι τροπολογίε. Ελπίζω να είναι επικοδομητικέ. Εγώ με, ανοιχ... ανοιχτό πνεύμα θα τι εξετάσω όλε. Ξέρετε, κάποιοι λένε. αν βέβαια πάρω τροπολογία η οποία θα μου λέει ότι πετάξτε όλα αυτά στα σκουπίδια που έχετε κάνει, ε, δεν θα τη δεχτώ, αλλά όλες τις άλλες θα τις συζητήσουμε.